Επίτροπε, αύριο 10.30 θα γίνει η ε, ψηφοφορία και τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Πατρίσια Τόγια για την κοινωνική οικονομία. Η συγγήτρια έχει το λόγο για 4 λεπτά. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ περήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την ε, κοινωνική οικονομία και θα αποφασίσει να ε, προωθήσει συγκεκριμένες προτάσεις για να υποστηρίξει αυτόν τον τομέα. Έχω τρεις σκοπούς να προωθήσω. Καταρχάς, να δοθεί προσοχή ε, για μια πολύ σημαντική πραγματικότητα που έχει και οικονομικό βάρος. Το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανήκουν σε αυτόν τον τομέα και το 9% των θέσεων απασχόληση. Μιλάμε για συνεταιρισμού, για ιδρύματα, για ενώσει ε, κοινωνική αλληλεγγύη, με συγκεκριμένε αξίε ε, που συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στο ΑΕΠ. Επομένω, θα πρέπει να δώσουμε μια θεσμική ορατότητα ε, πιο ξεκάθαρη. δεύτερο στόχο. Να τονίσουμε ότι αυτός τομέα δεν είναι ένα τομέα περιθωριοποιημένο, μια εξαίρεση, αλλά βρίσκεται ενταγμένο στην οικονομία τη αγορά, με του δικού του κανόνε. Ε, που θα πρέπει να αναγνωριστούν και να γίνουν σεβαστοί. Ένα διαφορετικό τρόπο για να παράγουμε, για να καταναλώνουμε, για να δίνουμε δουλειά. Ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί γιατί ανήκει στην οικονομία τη αγορά. Ε, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν θα πρέπει να τα ε, εξαλείψουμε. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε, λένε αυτές οι εταιρείε την αγορά, την απασχόληση, την παραγωγή και την κατανάλωση με την αξιοπρέπεια ε, του ανθρώπου. Ε, αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με το κεφάλαιο, αλλά όχι για το κεφάλαιο. Είναι τμήμα ε, της πραγματικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική οικοτομία είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αλλά εμείς τι κάναμε συγκεκριμένα. Είναι κατάλληλη στιγμή σήμερα για να ανακαλύψουμε την πραγματικότητα αυτών των επιχειρήσεων γιατί ε, η σημερινή κρίση έδειξε ότι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις συχνά είναι πολύ ε, ασταθείς, πολύ ευπαθείς. Αντίθετα, αυτή η οικονομία είναι συνδεδεμένη με την ε, τοπική πραγματικότητα, με, το, με, τα, με τους ανθρώπους και επομένως αντιστέκεται στις κερδοσκοπίες, αντιστέκεται γενικά. Επίσης, προωθεί η ευημερία του ανθρώπου, Προωθείται την κοινωνική αλληλεγγύη Επίσης ε, στηρίζονται σε, δύσκολε στιγμού, ε, δύσκολες στιγμές ε, τα κοινωνικά μας συστήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να υποστηρίξουμε αυτόν τον τομέα. Θα σας κάνω κάποιες προτάσεις πολύ σύντομα. Θα πρέπει καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμούς για να καταλάβουμε το προφίλ και το είδος του κάθε τέτοιου φορέα κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, θα πρέπει στους εθνικούς λογαριασμούς της κάθε χώρας να δούμε πόσο συνεισφέρει αυτός ο τομέας ε, δεν, είναι δημόσιοι οι φορείς αυτοί, δεν ανήκουν στην καπιταλιστική οικονομία. Ε, θα μπορούσαμε ε, η Κομισιόν να προωθήσει ένα εγχειρίδιο, ας πούμε, υπέρ αυτών των ε, ενώσεων. Νομίζω ότι ακόμη και τα πανεπιστήμια ε, και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Επίσης, χρειαζόμαστε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μπορεί να χρειάζονται. Ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε διαβουλεύσεις. Θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Δεν θέλουμε εμείς να οδηγήσουμε σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται, χρειάζονται και κοινοτικοί κανόνες. Έπειτα, ε, σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει μια έδρα ούτως ώστε να γίνει ένας διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, χρειαζόμαστε προγράμματα ad hoc ή θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την κοινωνική οικονομία στα σημερινά προγράμματα. Ας το αξιολογήσει αυτό η Κομισιόν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εθνικές ε, οργανώσεις, τα εθνικά δίκτυα που με πλαισίωσαν σε αυτή τη δουλειά. Την διακομματική οργάνωση του Κοινοβουλίου, ε, τους σκιώδεις εισηγητές και τον Επίτροπο. Σας δίνουμε αυτή την έκθεση, ε, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ε, οι κοινωνικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών και ελπίζω ότι παρά τις δύσκολες στιγμές θα βρείτε, κύριε Επίτροπε, το χρόνο μια και εκπροσωπείτε εσείς εδώ την, όλη την Επιτροπή, για να προωθήσετε μια κάποια πρωτοβουλία και για αυτή την κοινωνική οικοτομία ούτως ώστε η επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο να μην ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά από κάτι το συγκεκριμένο, κάτι το απτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Τόγια. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ευρωβουλευτέ, η Επιτροπή χαίρεται για την πρωτοβουλία, αυτή την ίδια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκπονήσει έκθεση όσον αφορά την κοινωνική οικονομία. Ιδιαίτερα σήμερα σε πλήρη οικονομική κρίση αξίζει πολύ μια τέτοια πρωτοβουλία. Όντω, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνει κανείς business. Μπορούμε δηλαδή να συνδυάσουμε την οικονομία με κοινωνικούς στόχους και να είναι αυτός ο επιχειρηματικός στόχος. Οπότε, όντως, ε, τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν και στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της υπαίθρου και της προστασίας του περιβάλλοντος, των καταναλωτών αλλά και της κοινωνικής ασφάλισης. Όντως, αποτελούν μέρος της πολιτικής για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επειδή οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εποφελούνται ήδη από το Small Business Act Στόχος μας όσον αφορά την κοινωνική οικονομία είναι να δημιουργήσουμε ένα νομικό και διοικητικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος όπου οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας υπό οποιαδήποτε μορφή ή μέγεθος να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ε, παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας μπορούν να μεγαλώσουν, να ευημερήσουν, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή για να φροντίσει και οι άλλες κοινωνικέ ε, πολιτικές, ε, είτε πρόκειται για το επιχειρηματικό δίκαιο, είτε πρόκειται για τις δημόσιες προμήθειες, για γεωργία, αλία, οι εταιρικέ σχέσεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα, όλες τις πάντων οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών, το ήθο, το είδο λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών κλπ. Εν κατακλείδη, υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπονούν έγγραφο το οποίο ε, σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2004 και μετά για την πρόθεση συνεταιρισμών και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και άλλων ε, τέτοιων επιχειρήσεων ε, κοινωνικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αύριο 10.30 θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Η μέληση διάταξη προβλέπει τώρα την έκθεση της κυρίας Ευαγγελίας Τζαμπάζη για την ψυχική υγεία. Παρακαλώ την εισηγήτρια, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει υγεία